παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, δέκα ημέρες μετά τον τυφώνα Χαϊάν που σάρωσε με πάνω από 300 χιλιόμετρα ολόκληρες εκτάσεις της Φιλιππίνης για εκατοντάδες χιλιάδες επιζώντες παραμένει δραματική η κατάσταση. Γνωρίζετε όλοι τις εικόνες ε, απελπισμένων ανθρώπων που δεν έχουν πόσιμο νερό, καθόλου φαγητό και είναι υποχρεωμένοι να διεκτερεύουν στην Ήπεθρο. Έχει αρχίσει να φτάνει η βοήθεια, αλλά παραμένουν ορισμένες περιφέρειες αποκομμένες από τον έξω κόσμο. Είναι ε, περίγραπτο το χάος που επίκρατει εκεί. Ε, Βοήθεια και τα συνεργεία διάσωσης ε, ε, αναζητούν αγνοωμένους, αγωνίζονται μέσα στα συντρίμια, άνθρωποι να επιβιώσουν και χρειάζεται βοήθεια διεθνής από το εξωτερικό. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να βοηθήσει τον κόσμο αυτό όσο ε, γίνεται πιο γρήγορα που το έχει τεράστια ανάγκη και για την ανοικοδόμηση των χωριών και των πόλεων που έχουν καταστραφεί χρειάζεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, δίνει και επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και πιο μακροπρόθεσμη έχει δεσμευτεί αλλά νομίζω ότι μπορούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε περισσότερα είναι δραματική η κατάσταση 11 εκατομμύρια άνθρωποι στις Φιλιππίνες ε, πλήττονται από τις συνέπειες αυτού του τρομακτικού τυφώνα. Είναι δραματικά τα αριθμητικά στοιχεία. 660.000 άνθρωποι είναι άστεγοι, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και σύμφωνα με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό είναι ακόμα 22.000 οι αγνοούμενοι, ενώ ο αριθμός των νεκρών θα το διαβάσατε, είναι πάνω από 2.500. Οι ε, οργανώσεις βοηθείας μας λέγουν ωστόσο ότι τα ε, στοιχεία αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν οπωσδήποτε. Θα ήθελα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απευθυνθώ στους πληγέντες και να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ε, ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση και σίγουρα Είμαι βέβαιος ότι ε, μοιράζετε κι εσείς μαζί μου τα αισθήματα της αλληλεγγύης ε, με τις οικογένειες και τα θύματα. Και θα σας παρακαλούσα να τηρήσουμε ενός λεπτού ε, σιγή. Και σας παρακαλώ να γερθείτε από τις θέσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να καλωσορίζω 150 μαθητές και μαθήτριες από 33 ε, χώρες. Καλωσορίσατε στη Euroscola. Είναι μια διημερίδα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά